ιδιωτικός με περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε. Τώρα συνάδελφοι θα αρχίσουμε το επόμενο θέμα μαζί με την ΑΝΑΦ, την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το Frontex. Στην έκθεση του του 12 ο διαμεσολαβητής είχε μιλήσει για την συμμόρφωση του Frontex προς το σεβασμό των φεμελιωδών δικαιωμάτων. Την ενέκρινε εκτός από ένα σημείο που αφορούσε την εφαρμογή της διαδικασίας προσφυγών για παραβίαση των, των βασικών δικαιωμάτων. Ο διαμεσολαβητής λοιπόν ζήτησε τη στήριξη του Κοινοβουλίου γι' αυτό. Η έκθεση του Κοινοβουλίου μετά από συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών ετοιμάστηκε από δύο συζητές, την κυρία Κέλλερ και την κυρία Μετσόλα. Σήμερα θα συζητήσουμε την έκθεση αυτή, οι συντονιστές συμφώνησαν η διορία κατάθεση τροπολογιών να λύγει αύριο 11 Νοεμβρίου στις 12. Η εξέταση των τροπολογιών προβλέπεται για τις 12 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 16 Νοεμβρίου. Το χρονοδιάγραμμα επιταχύνθηκε για να μπορέσει να υπάρξει θέση του Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια πριν την κατάθεση νέων προτάσεων από την Κομισιόν για το νομικό του Frontex. Έχουμε εδώ μία αντιπροσωπεία του Frontex και του διαμεσολαβητή για να απαντήσουν σε πιθανές σας ερωτήσεις. Δίνω πρώτα το λόγο στη συνάδελφό μου κυρία Βίκστρομ, πρόεδρο της Επιτροπής ΑΝΑΦ και μετά στους εισηγητές και ύστερα στους υπόλοιπους. Ορίστε κυρία Βίξτρομ μου. Ευχαριστώ κυρία Ιώτοβα. Και εγώ σας καλωσορίζω σε αυτή την κοινή συνάντηση με τη Λίμπε ως πρόεδρος της Επιτροπής ΑΝΑΦ. Όπως είπε μόλις η κυρία Ιώτοβα είναι η πρώτη τέτοια κοινή συνάντηση για τη συζήτηση αυτού του σχεδίου έκθεση. Επίσης ευχαριστώ την προσοχή στο γεγονό ότι και το Frontex και το γραφείο του διαμεσολαβητή αντιπροσωπεύονται σήμερα εδώ, εκπροσωπούνται. Από το Frontex έχουμε τον κύριο Τζι Λαρίας, τον διευθυντή του και τον κύριο Ευρέ Κανιάρ. Και από τον διαμεσολαβητή η Μάρθα Χίρς, Σεμπίνσκα, τμήματάρχης. Παρακαλώ να θέσετε όσες ερωτήσεις θέλετε. Καταρχήν, να αρχίσει η συζήτηση με τους εισηγητάς, την κυρία Μετσόλα και την κυρία Κέλλερ. Θέλετε να αρχίσετε εσείς κυρία Κέλλερ. Ναι, η συνεργασία με τον, την συνεισηγήτριά μου κυρία Μετσόλα ήταν εξαιρετική. συνεννοηθήκαμε μεταξύ σκιωδών. Δεν θα υπησέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά να σας πω μόνο γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει τέτοια διαδικασία προσφυγών και παραπώνων. για όσους δηλαδή θεωρούν ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους στα πλαίσια μιας επιχείρησης του Frontex. Αυτό συζητιέται στα πλαίσια του νέου ρόλου του Frontex στα hot που η Κομισιόν προβλέπει να καταθέσει νέες προτάσεις ήδη τον επόμενο μήνα. Επίσης δεν υπάρχει νομικός φραγμός για να δημιουργηθεί μια τέτοια διαδικασία. Όσοι θεωρούν ότι έχουν βλαφθεί τα δικαιώματά των, πρέπει να μπορούν να προσφεύγουν. Ιδίως για περιπτώσεις που χωρίς την προσφυγή δεν θα γινόταν γνωστό το πρόβλημα. Τώρα ο μηχανισμός που προτείνεται είδαμε πρώτα το υπάρχον εσωτερικό σύστημα πληροφόρησης που διαθέτει το Frontex υπάρχει και ιδιωκός αξιωματούχος για τα θέματα παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που, τον οποίο είχε προβλέψει ήδη το Frontex από πριν. Ο μηχανισμός προσφυγής ή παραπώνων θέλουμε να είναι αποτελεσματικό κος να αφορά και μη κυβερνητικές οργανώσεις και την υποβολή του παραπώνου στις γλώσσες που μιλούν οι ενδιαφερόμενοι. Βεβαίως στα πλαίσια του Frontex αυτό θα σήμαινε ότι χρειάζονται ειδικοί καινούργοι αξιωματούχοι γιατί το Frontex δεν έχει ειδική διακοδοσία για αυτό το θέμα. Γι' αυτό συνήθως μέχρι σήμερα τα μετέφερε τα παράπονα σε εθνικές αρχές. Εμείς θέλουμε το, η χώρα μέλος που θα λάβει τέτοια προσφυγή να την διεκπαιρεώσει πράγματι. Επίσης μπορεί να κάνει κάτι και το ίδιο το Frontex ας πούμε να αποκλείσει όποιον αξιωματούχο του έχει παραβιάσει θεμελιώδη δικαιώματα από βασικές επιχειρήσεις του να αποσύρει χρηματική βοήθεια από κράτη-μέλη που δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα παράπονα και μετά την τελευταία του, με την τελευταία μορφή της εντολής του να μπορεί να σταματήσει, να τερματίσει μια επιχείρηση αν έχουν διαπιστωθεί παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχουν λοιπόν θέματα που μπορεί να λύσει και μόνο του το Frontex όσο για τους λεγόμενους guest officers θα μπορούσε ο μηχανισμός αυτός να γίνει σεβαστός με βάση τις ε, προτάσεις του διαμεσολαβητού. Βεβαίως αν υπάρξει ένας τέτοιος καινούργιος ηθικός αξιωματούχος πρέπει να έχει και τα, μέσα, τα χρηματικά μέσα για να ανταποκριθεί στην εντολή του. Ευχαριστώ ξανά τους Κιώδης και υπενθυμίζω ότι η διορία λύγει αύριο στις 12 για τις ντροπολογίες. Ευχαριστώ ξανά την κυρία Μέτσολα. Ευχαριστούμε κυρία Μέλλερ και τώρα η κυρία Μέτσολα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για την συνεργασία. Σύνταξαμε μαζί το κείμενο σε σχέση με την έκθεση του Δημοσιολαβήτη και την Frontex. Ευχαριστούμε επομένω όλους τους και οδησίδες. Με την πρόεδρο στην Επιτροπή Αναφορών και την εκπροσωπώ βεβαίως, όσον αφορά το ζήτημα. Και έχουμε στο κείμενο ε, την τοποθετησή μας, δηλαδή είμαστε υπέρ της υποστήριξης της ε, Frontex, λάβουμε υπόψη τα όσα περισσεύει το Κοινοβούλιο για την ε, Frontex και είπαμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο μηχανισμός υποβολής εκθέσεων και κοινοποίησεων και επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα γραφείο θεμελιών δικαιωμάτων στην ε, Frontex. Αλλά βέβαια να ε, ε, την χάνει ανεξαρτησίας. Επίσης θεωρούμε ότι η Frontex μπορεί να εξασφαλίσει την περιφρούρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί να χειριστεί και τον μηχανισμό των ατομικών καταγγελιών. Δεν θέλουμε να παραβλάσουμε την έκθεση αυτή τη αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε των κρατών μελών. Να σεβαστούμε την αρχή τη επικουρικότητα. Και ρητό λέμε στο κείμενο ότι η Frontex δεν έχει αρμοδιότητα να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο ε, σε πρόσωπα πέραν του προσωπικού της Frontex. Ο κανονισμός της Frontex είναι σαφής. Πειθαρχικά μέτρα είναι θέμα κρατών μελών, κρατών μελών προέλευσης. Πάντως έχουμε και αυτό το μηχανισμό για τις ατομικές καταγγελίες. Οπότε ο κόσμος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του για ε, ε, να προσφύγει στη δικαιοσύνη με τελεσματικό τρόπο. Σε περίπτωση παραβίασης ε, θύμιλων δικαιωμάτων και θέλουμε έτσι να καλύψουμε κάποιες περιπτώσεις που δεν θα καλύπτονται από άλλου είδους διατάξεις οπότε θεωρούμε ότι τώρα υπάρχουν όλες οι εγγύσεις για να έχουμε την κάλυψη όλων των περιπτώσεων παραβίασης δικαιωμάτων και των σχετικών τους ε, ε, καταγγελιών. Βέβαια καλύπτονται εδώ τα δικαιώματα που υπάρχουν στον χάρτη των θεμελιωτών δικαιωμάτων, μόνο αυτά τα δικαιώματα. Και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα να παράσχουν ε, ό,τι πόρου χρειάζεται η Frontex, ούτω ώστε να μπορούσε η Frontex να ασκήσει ε, αυτέ τι αρμοδιότητε σε σχέση με αυτά τα δικαιώματα με αποτελεσματικό τρόπο. Περιμένω να ακούσω τι προτάσει σα συνάδελφοι αλλά και από τους σχεδόν Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους ε, Κέλ και Μετσόλα για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Ε, πραγματικά είναι μεγάλη ικανοποίηση που ε, αυτό το κοινοβούλιο στην ουσία ανταποκρίνεται στη δουλειά που έχει κάνει ο διαμεσολαβητής. Να σας δώσω κάποια στοιχεία σχετικά με την σημασία αυτού του θέματος. Τα τελευταία χρόνια, καταρχάς, έγιναν πολλά βήματα για να διασφαλίσουμε ότι η Frontex θα είναι ο μηχανισμός που θα διασφαλίζει την συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και Φυσικά οι κανόνες για τα θαλάσσια σύνορα ήταν μεταξύ αυτών των ε, προόδων. Βέβαια, ε, ε, υπάρχει αυτή η ρύθμιση στα επιχειρησιακά σχέδια να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Υπάρχει μια σειρά υποχρεώσεων και ευθυνών για την Frontex και τους ε, αξιωματούχους που συντονίζει. Στο προσεχές ε, μέλλον θέλουμε να αυξηθεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θα επηρεάσει και τη Frontex γιατί το πεδίο δράση της έχει να κάνει ακριβώς με τη συμμόρφωση με αυτό τον κανονισμό και όχι με τα κράτη-μέλη. Ο ρόλος τώρα της Frontex είναι ξεκάθαρο ότι ο ρόλος αυτός ε, αλλάζει συνεχώς, ε, όμως ε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι χρειάζονται περισσότεροι ελεγκτικοί μηχανισμοί και για τους πολίτες για να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα και όλες τις επιχειρήσεις της Frontex. Τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί το πεδίο δράσης της Frontex, αλλά και τα μέτρα για το σεβασμό των δεμελιωδών δικαιωμάτων. Το μέλλον θα πρέπει να ακολουθήσει τα ίδια βήματα. Ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Μίλνε. Παρακαλώ σεβαστείτε το περιθώριο των δύο λεπτών, γιατί δεν έχουμε χρόνο και είναι νέα συνόλφοι που θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Θα σεβαστώ σίγουρα τα δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές τι δύο συγκίτρε, μάλλον, την κυρία Ματσόλα και η Κέλνερ για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν. Είναι πολύ καλό το συμβαστικό κείμενο. Ναι. Ειλικρινά θεωρώ ότι εδώ υπάρχει ένας καλός μηχανισμός ε, για τις προσφυγές σε περίπτωση παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι βασικό επίτευγμα του Κοινοβουλίου. Μέσα στα πλαίσια του τρέχοντος κανονισμού για τη Frontex, ε, η διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, δεν ε, έχει την, την απαραίτητη ε, θέση, πρέπει να βελτιωθεί στους επόμενους κανονισμούς όσον αφορά στην πολιτική επιστροφή σε έρευνα και διάσωση. Ο μηχανισμός πρέπει να είναι δίκαιος, να λαμβάνει υπόψη την ευαίσθητη κατάσταση των μεταναστών και του τον αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι και ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος. Θεωρώ ότι είναι καλός συμβασμός, αλλά χρειάζονται και κάποιες προσαρμογές κατά τη γνώμη μου. Χρειάζεται ένα follow-up, ένας μηχανισμός αναφοράς για τις ε, προσφυγές. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ της Frontex και των Οργανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Και τέλος, αλλά όχι εσχάτως, χρειαζόμαστε και η ημερήσια διάταξη να είναι ε, ευαίσθητη σε θέματα φύλου ε, και τα λοιπά. Συχνά οι άντρες ενημερώνονται μόνο και όχι οι γυναίκες για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, για τα δικαιώματα προσφυγής ε, σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Thank you. And the next, uh, Madame... Ευχαριστώ η κυρία Ρουίς. Sí, muchas gracias. Ε, κυρία, Καταρχάς ε, θα ήθελα να συγχαρώ τις εισηγήτριες. Είναι πάρα πολύ ε, επενέντα αυτό το οποίο λένε, αλλά θέλω να δούμε και κάτι άλλο. Πέρα από αυτούς τους μηχανισμούς που περιέχει το σχέδιο κειμένου, το οποίο μου φαίνεται βέβαια κατά τα άλλα πολύ καλό, τι γίνεται για την μη ενημέρωση κάποιων ομάδων ευάλωτων. Και μιλώ για κάποιες ομάδες που βρίσκονται εκεί που δράει η Frontex και που ε, τα δικαιώματά τους. Ιδίως οι μη συνοδευόμενοι ανήλικοι κάποιοι ΛΟΑΔ, κάποιοι ηλικιωμένοι. Όλοι αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά του τα οποία παραβιάζονται. Θα πρέπει ομένως να γίνει η επισήμανση αυτών των ευάλωτων ομάδων και να υπάρχει κάποια πολύ συγκεκριμένη πρόβλεψη για αυτές τις ομάδες. Κύριος Κύρχοπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε λίγο χρόνο, απλώς να πω ότι η ομάδα μου υποστηρίζει τους συνολικούς στόχους σχετικά με τη διαδικασία προσφυγών. Έχω ένα-δύο ερωτήματα όμως. Θέλω να μάθω πώς γίνεται το follow-up των προσφυγών. Γιατί η κατάσταση των προσφύγων ε, μπορεί να είναι μεταβατική, δεν υπάρχουν ένδικα μέσα που να είναι δυνατά, ε, πώς μπορούν να δοθούν οι νομικές συμβουλές ε, στους προσφεύγοντες. Τι ακριβώς είναι αυτό που καθιστά παραβίαση των ε, θεμελιώδων δικαιωμάτων. Είναι ένα κοινό κριτήριο ή το κάθε κρατός μέλος έχει τα δικά του κριτήρια ή τα ερμηνεύει όπως θέλει. Ποια είναι η διαδικασία για άλλα, άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί η δουλειά της Frontex είναι τελείως διαφορετική και θεωρώ ότι οι διαδικασίες αυτές ε, ως έχουν ε, δεν θα είναι αποτελεσματικές για τη Frontex σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κύρκοπ και τώρα θα δώσω το λόγο στους σκιώδης Η Κυρία Καλή έχει το λόγο πρώτη. Thank you, ε, Definitely. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως ε, η αντιμετώπιση των αδυναμιών είναι σημαντικό στοιχείο και γι' αυτό η ομάδα μου, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, όντως υποστηρίζουν ε, αυτό το αίτημα του δημιουργίας μηχανισμού προσφυγών για, τα... για το θέμα της τραβής των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τίποτα βέβαια στον τρέχοντα κανονισμό δεν εμποδίζει τη Frontex να κάνει ένα τέτοιο μηχανισμό. Η διάσωση σώων είναι η προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο με ανησυχεί το πώς ακριβώς ορίζεται η η επιχείρηση διάσωσης ζωών. Αυτό μπορεί να αντιβαίνει στα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε μηχανισμός υπάρξει δεν θα αποτρέψει, δεν θα σταματήσει, δεν θα επηρεάσει τη διαδικασία ασύλου, γιατί πρέπει τις καταχρήσεις να αντιμετωπίσουμε. Μετά, η, διαβα... η διαφάνεια είναι πολύ ζωτική σημασία σε αυτή τη διαδικασία. Η ομάδα μου λοιπόν προτείνει η Frontex να έχει μια ετήσια έκθεση που θα περιλαμβάνει πληροφορίες ε, για τις προσφυγές που έχουν γίνει και το follow-up. Το να κατανοήσουμε ποια είναι τα ε, αιτήματα, ποιες είναι οι προσφυγές ε, και ποια τα μέτρα θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το πεδίο εφαρμογής ε, και νομίζω ότι τα, οι οργανισμοί θεμελιωδών δικαιωμάτων θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Τρίτον, Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αξιωματούχοι για τα θεμελιώδη δικαιώματα παίρνουν περισσότερη υποστήριξη. Δεν είναι θέμα μόνο οικονομικής βοήθειας. Ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε από μια τόσο μικρή ομάδα να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο έργο. Περιμένουμε περισσότερα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αξιωματούχοι αυτοί έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουν να επιφέρουν περισσότερα αποτελέσματα. Τέλος, πρέπει να διασφαλίσουμε τις ε, ευαίσθητες ομάδες όπως τους ε, ασυνόδευτους ανήλικους ε, μέσα από ε, συνεργασία με την ΕΑΖΟ και παρόμοιους οργανισμούς. Συν... Τελειώνοντας να πω ότι προσβλέπουμε στη συνεργασία με τους εισηγητές για αυτό το θέμα. Ο κύριος Νάγκη είναι ο σκιώδης εισηγητής και όχι η κυρία Νταλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την λεπτομερή εργασία των εισηγητών. Το ΕΛΚ υποστηρίζει πλήρως ε, το μηχανισμό προσφυγών ε, ως προς τη δουλειά της Frontex. Ε, σύντομα να πω ότι θεωρώ πως είναι ανάγκη να τονίσουμε τον... την ανάγκη να μην θέσει περισσότερο διοικητικό φόρτο και νέες ευθύνε στη Frontex ο νέος μηχανισμός. Επίσης πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της συμμόρφωσης των τρίτων μερών σε αυτό τον ε, μηχανισμό. Τέλος, ε, να μιλήσουμε και για τις δυνατότητες των ανθρώπων που μπορεί να χρειάζονται βοήθεια για να συμμορφωθούν. Τώρα θα δούμε ποιες θα είναι οι τροπολογίες και θα δούμε και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Ευχαριστούμε και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Τζουάρτ Μαρτά από την Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συγχαίρω και εγώ τους δύο εισηγητές. Όλοι συμφωνούν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει αυτή η νομοθεσία, η ρύθμιση. Καταθέσουμε και εμείς ορισμένες τροπολογίες. Βασικά όμως είναι μια καλή, καλό σχέδιο έκθεσης για να υπάρξει καλύτερη εγγύηση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συνδυάζει σωστά το Frontex με τις κρατικές εθνικές υπηρεσίες. Εμείς θα ζητήσουμε κάπως καλύτερη νομοθεσία για τους πιο ευάλωτους γυναίκες, παιδιά. Απ' την άλλη όμως, για μας αποκλείεται να απορρίψουμε τις ανώνυμες προσφυγές. Γιατί πολλές φορές η ανωνυμία οφείλεται σε πολύ σοβαρά ως λόγους. Πρέπει να τις δεχτούμε λοιπόν και αυτές. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μαρτέν. Η κυρία Μπιόρκα από την Επιτροπή ΕΛΕΦ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ εκ μέρους της ομάδας μου χαιρετίζω το γεγονός ότι θα υπάρξει ένας τέτοιος ε, μηχανισμός ε, γιατί υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και είναι σημαντικό να δοθεί η ιδέουσα σημασία στη δουλειά της Frontex Εδώ ε, στην έκθεση πρέπει να δώσουμε σημασία στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έδωσαν τα φώτα τους. Ε, μια πρόταση για ένα πιλωτικό λοιπόν έργο να ενισχυθεί αυτή η εργασία είναι καλή. Ένα όμως βασικό πρόβλημα υπάρχει με μας. Ο μηχανισμός προσφύγων πρέπει να μπει στο πλαίσιο της Frontex δεν ε, γίνεται να περάσει αυτός ο μηχανισμός ε, εντός της Frontex, ε, πρέπει να είναι εκτός Frontex και γι' αυτό οι υπάλληλοι των, της Frontex και των κρατών μελών αλλά και το προσωπικό των τρίτων χωρών πρέπει να ληφθούν υπόψη. Νομίζω λοιπόν ότι όταν υπάρχει μια παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανώνυμης ε, καταγγελίας ε, για να μπορούμε να έχουμε και την ισότητα που επιθυμούμε για τις γυναίκες, για παράδειγμα. Πρέπει και αυτές να ληφθούν υπόψη και τρίτον και τρίτη, θα μπορούν επίσης να καταθέτουν ας πούμε μία προσφυγή, για παράδειγμα οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Τώρα, μετά τους κοιόδες, θα δώσω το λόγο στην κυρία Λάουρα Φεράρα, μετά στην κυρία Γκοσμάν και μετά θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μουσουλίνη. Μετά κλείνει ο κατάλογος. Euh, Κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια και από μένα στις δύο συντάκτριες και για τον διαμεσολαβητή για αυτήν την ε, έρευνα μια που ανταποκρινόταν στο ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και από φυσικά πρόσωπα. Οπότε τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τους ε, μετανάστες αυτό αυτό το οποίο ήταν σημαντικό και έλειπε. Οπότε αυτό το οποίο για μας έχει σημασία και θα πρέπει να αναδείξουμε είναι το ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον εσωτερικό μηχανισμό ε, δεν, που ε, θα πρέπει να έχει όλες τις ε, εγγύσεις της ανεξαρτησίας. Θα πρέπει να υπάρχει μια ανάλυση αντικειμενική σε σχέση με τις καταγγελίες. Οπότε γι' αυτό και για να βελτιωθούν οι εγγύσεις αυτές, εμείς προτείνουμε με τροπολογίες ένα πάνελ εξωτερικών συμβούλων που θα εγγυηθούν την ανεξαρτησία και για οι καταγγελίες που θα πρέπει να αφορούν μόνο τις σοβαρές παραβιάσεις. Εμείς ε, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να θεωρούνται για τυπικούς λόγους οι καταγγελίες ε, απαράδεκτες και οπότε θα πρέπει πέραν των τυπικοτήτων να εξετάζεται πάντοτε η ουσία της καταγγελίας. Επομένως θα πρέπει να δούμε ε, ποιες είναι σοβαρές καταγγελίες και ποιες όχι, αλλά να υπάρχει έτσι η δυνατότητα για πάσα καταγγελία να ασκείται. Ε, κάπου εκεί που κατοχυρώνεται η, η ανωνυμία του καταγγέλλοντος είναι ένα άλλο σημείο. Θα πρέπει και εδώ να υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις και έτσι να αποφύγουμε κάποιος από φόβο να μην καταγγέλει. Είναι σημαντικό το θέμα της ε, πληροφόρησης και για τους ετούντες άσυλο και για αυτούς που εκεί εργάζονται. Ε, άρα σε όλες τις γλώσσες να υπάρχει ενημέρωση, σε όλες τις γλώσσες ε, στις οποίες μιλούν οι μετανάστες. Ευχαριστούμε κύριε Φεραλία Πρόεδρος για τώρα ε, το λόγο η κυρία Γκούσμαν. Σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε τις δύο συντάκτριες. Μιλούμε τώρα για τη φρόντιση και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Άρα το πρώτο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι πώς θα γίνει ο έλεγχος της μεθορίου. Να γίνεται χωρίς παραβίαση δικαιωμάτων ε, πρώτα-πρώτα ε, ε, πάρα πολλοί που ρισκάρουν την ζωή τους στη θέωτα, τη μελίγια, στη θάλασσα θαλασσοπνίγονται και προσοχή να μην κινδυνεύουν περισσότερο από τον έλεγχο η Frontex έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο των συνόρων και όχι τίποτε άλλο, άρα να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα. Επίσης ε, να προσέξουμε κάποιες πρακτικές ε, που κάνουν τα πράγματα πιο ε, σοβαρά και οπότε γι' αυτό και ο διαμεσολαβητής τώρα στην προσοχή του για κάποιες μακρές πτήσεις που αφορούν κάποιους επαναπατρισμούς, μεταφορά προσφύγων τι γίνεται ας πούμε για κάποιο είδους ε, πλωτά μέσα πάνε στην, ε, ε, πάνε στη Λέσβο και προσπαθούν να σώσουν αυτούς τους 300 επιβάτες έτσι μας είπε ένας εθελοντής και θα πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός για καταγγελίες εκεί στα σύνορα οπότε θα πρέπει να λέμε να διαλυθεί η φρόντες, να σταματήσουν οι, οι επάνθρωπες πρακτικές και να σταματήσουν επίσης και οι απελάσεις. Έτσι να έχουμε περισσότερη διαφάνεια και θα πρέπει να υπάρχει περισσότερους περισσότερος έλεγχος όσον αφορά τη Frontex. Λοιπόν, θα πρέπει όλες οι διαδικασίες να είναι ε, δημόσιες, όλα να καλύπτουν τον προϋπολογισμό και να υπάρχει έλεγχο κοινοβουλευτικό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε προ αυτέ τι κατευθύνσει τροπολογίε που θα υποβάλουμε. Θα λέω, είναι η τελευταία που θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μόνο μία ερώτηση έχω που έχει να κάνει με τους απεσταλμένους υπαλλήλους συγκεκριμένα αυτές οι πειθαρχικές διαδικασίες μπορούν να εφαρμοστούν όταν ε, ε, συνενέσει το κράτος μέλος. Ε, εντάξει, ίσως αυτό να αρκεί, δεν μπορώ να πω κάποια άποψη γι' αυτό. Ίσως αργότερα να μπορεί να αλλάξει βέβαια. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει τα κράτη-μέλη αυτά τα ίδια να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως τα δικαιώματα των παιδιών και τα λοιπά και αυτοί που αποστέλλονται ως υπάλληλοι να έχουν μια καλή βασική εκπαίδευση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Όταν λοιπόν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές τελικά για το πώς αντιμετωπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε πρέπει να ε, διαμορφώσουμε κάπως αλλιώς το σύστημα στο μέλλον, ενδεχομένως. Ευχαριστώ το λόγο, κύριε. έχει, έχει η κυρία Μουσολίνη. Εγώ, Πρόεδρε, θα θίξω ένα σημείο, γιατί κατά τα λοιπά συμφωνώ για αυτούς τους ευάλωτους και κυρίως όσον αφορά τους κινδύνους και τα δικαιώματα των ανηλίκων. Και θέλω επίσης και εγώ να συγχαρώ τις ε, συντάκτες που θέλουν να αποκτήσει ανθρώπινο πρόσωπο η Frontex, μια από τώρα ε, επιτελεί τόσο σημαντικό ρόλο. Γιατί είναι και κάτι άλλο. Θα πρέπει να δούμε και να διεκδικήσουμε πώς θα γίνει η διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να σταματήσουν οι παραβιάσεις. Και θα ήθελα να αναφερθώ στις καταγγελίες θα πρέπει πέραν τον άλλον να δούμε τι γίνεται στην πραγματικότητα και στην Ιταλία και αλλού. Δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα αυτοί οι μετανάστες. Κάποιοι έχουν διαβατήριο και κάποιοι έχουν ε, ταυτότητα, δεν έχουν έγγραφα οι περισσότεροι. Οπότε τελικά οι καταγγελίες που γίνονται είναι ανώνυμες για αυτό το λόγο. Όμως δεν μπορεί να γίνει η Frontex ένα δικαστήριο. Θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητες που έχει, όπως το λέει και το κείμενο. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με εκείνους τους μετανάστες που δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα ή άλλα έγγραφα και που είναι το μεγαλύτερο μέρος αυτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόμπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σχεδόν λαμβάνεται ως δεδομένο ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι μας, θα υποστηρίξουμε τη δέσμευση της Frontex στα θεμελιώδη δικαιώματα. Το σημαντικό όμως είναι ότι ήδη έχει αναθεωρηθεί η εντολή της Frontex ακριβώς για να διασφαλιστεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχει ένας ειδικός ε, συντάκτης εντός ε, της Frontex, ε, μια ειδική μονάδα εντός της Frontex για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οπότε αναρωτιέμαι ποια ήταν ε, η ουσία της αναθεώρησης της εντολής της Frontex το 6 και το 11 αν δεν κάνω λάθος ακριβώς για να ενισχυθεί αυτή η δέσμευση. Και δεύτερον, ποια είναι ακριβώς τα θεμελιώδη δικαιώματα που φέρεται, φέρονται ως τα πιο ε, συχνά ας πούμε θύματα παραβίασης. Ακριβώς ποια είναι λοιπόν αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναφέρονται στις αναφορές που έχουν γίνει ως τώρα και που γνωρίζουμε. Είναι θέμα γεγονότων. Θέλουμε να μάθουμε πιο συγκεκριμένα γεγονότα δηλαδή. Ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, έχουμε τρία λεπτά για δύο ομιλητές. Η κυρία Σπινέλη και τέλος η κυρία Γνόντα Λάνς. Ευχαριστούμε την Σκιώδη συγκίτρια και την συγκίτρια Πρόεδρε Δύο θέλω να αναφέρω δύο θέματα. Πρώτα πρώτα κάτι νόμο είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε το δικαίωμα προσφυγής των μεταναστών, να το αναφέρουμε στην έκθεση και ιδίω σε σχέση με τις ασφαλείς χώρες όπως τα είπε πριν από μένα νομίζω η κυρία Λάουρα Φεράρα. Και τώρα κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον θα πρέπει να μπει στην έκθεση. Θα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 263 της συνθήκης. Λέει ότι το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ασκεί έλεγχο νομιμότητος όσον αφορά τα όργανα και τις υπηρεσίες της Ένωσης που οι αποφάσεις τους ε, και έναντι τρίτων παράγουν νομικά αποτελέσματα. Αυτό για να τηρηθεί η δημοκρατική αρχή, αυτό το συνταγματικό δικαίωμα ε, προστασίας των πολιτών. Ευχαριστούμε κύριε Σπινέλη, λέει Πρόεδρος. Κύριε Ευχαριστώ. Υποστηρίζω πλήρως την δημιουργία αυτού του μηχανισμού προσφυγών που πρέπει να ισχύει και για επιχειρήσεις μέσα και έξω στην Ένωση. Υπάρχουν οι working agreements μεταξύ Frontex και τρίτων χωρών. Ο ε, βασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων ισχύει φυσικά και για το Frontex μέσα στις σχέσεις εργασίας του. Εφόσον μάλιστα δράει εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σεβασμός λοιπόν των θεμελιωδών δικαιωμάτων ισχύει και για τους πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά σήμερα δεν είναι υποχρεωτικός, δεσμευτικός πρέπει να γίνει και μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου γιατί έτσι θα ενδυναμωθεί η νομική ασφάλεια που μας λείπει εδώ. Η επέκταση λοιπόν του μηχανισμού αυτού και στις σχέσεις εργασίας θα δημιουργήσει μεγαλύτερη διαφάνεια γιατί αλλιώς δεν θα γίνονται καν γνωστές οι παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων μεταξύ άλλων και των μεταναστών και προσφύγων. Έχω καταθέσει σχετικό τροπολογίες, σας κατευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχουμε εδώ και δύο αντιπροσωπείες του διαμεσολαβητού και του φροντέρας. Μήπως θέλει κανείς από αυτούς να λάβει τον λόγο. Δίνω το λόγο πρώτα στο φροντέρας. Ποιος είναι, ποιος. Ποιος, εσείς κύριε μου. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση μου. Θέλω να σχολιάσω μερικά θέματα που αναφέρθηκαν από πολλούς βουλευτάς. Πρώτον, κατά πόσον το υπάρχον νομικό πλαίσιο αρκεί για να συσταθεί ένας επίσημος μηχανισμός προσφυγών ή παραπώνων. Δεν, δεν θα το συζητήσω αυτό, αλλά να τονίσω ότι με το υπάρχον νομικό πλαίσιο το σύστημα δεν είναι δεσμευτικό για τα κράτη-μέλη και άρα μπορούν να αποφασίσουν να συνεργαστούν ή όχι. Και απ' την άλλη εμείς δεν μπορούμε με την εντολή που έχουμε τώρα να διαχειριστούμε τα προσωπικά στοιχεία των παραπονουμένων μόνον για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις δουλεμπόρων ή λαθρεμπόρων. Για τις ανώνυμες προσφυγές. Αν το θέμα είναι η προστασία της ανωνυμίας του προσφεύγοντος τότε μπορούμε να το κάνουμε. Αν όμως εννοείται την διεκπαιρέωση ανωνύμων παραπώνων, τότε όχι δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Ε, concerning the individual complaints... Για ατομικές προσφυγές από το 2013 έχουμε λάβει μόνο τέσσερις και οι περισσότερες από αυτές ε, και οι περισσότερες για pushbacks, για pushbacks δεν έχουμε καταγράψει καμία παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων από guest officers. Δηλώσεις μεταναστών αφορούν κυρίως εθνικούς αξιωματούχους κατά τη διαδικασία επιστροφής σε χώρες, στις χώρες προέλευσης τους. Αυτά λέμε pushbacks, αυτό εννοούμε pushbacks. Αν έχετε, αν θέλετε περισσότερες εξηγήσει να μου πείτε. Ευχαριστώ. Τελευταία κυρία Τζιμπίνσκα, που εκπροσωπεί τον διαμεσολαβητή. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος του διαμεσολαβητού θα ήθελα να πω μερικά λόγια κι εγώ. Πρώτον, η ειδική έκθεση του Ombudsman είχε γραφτεί υπό το προηγούμενο καθεστώς του Frontex. Με το καινούριο το Frontex θα έχει περισσότερη αυτονομία στην ειδική έκθεση λέγαμε και στο σχέδιο έκθεση του Κοινοβουλίου ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και το Γενικό Δίκτυο Διαμεσολαβητών και Διαμεσολαβητριών θα συνεργαστούν με το Frontex όσο περισσότερο γίνεται με βάση την εμπειρία μας για τη διεκπαιρέωση παραπώνων και προσφυγών. Και από τα ερωτήματα που ακούστηκαν, τις ερωτήσεις για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό, με ποιο μηχανισμό κτλ. Ποιος θα ασχοληθεί ακριβώς. Εμείς μπορούμε να βρούμε, να δώσουμε λύσεις με βάση την εμπειρία μας, expertise. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στα πλαίσια των δικαιοδοσιών του διαμεσολαβητού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τζιμπίνσκα. Μήπως θέλουν και οι δύο εισηγητές το λόγο. Πόσο χρόνο έχουμε. Μείον 7 λεπτά. Ωραία. Θα είμαι λοιπόν σύντομη. Ευχαριστώ τους πάντες και τις πάσες για όσα είπαν. Ίσως γενικό σχόλιο θα έλεγα ότι είχαμε τη φοβερή πρόκληση να διασφαλίσουμε ότι θα μείνουμε μέσα στο πλαίσιο των των κανόνων του Frontex χωρίς να μπούμε στην υποθετική περίπτωση της αναθεώρησης των κανόνων του Frontex. Επομένως, θα δίναμε την ευκαιρία στο Frontex απλώς να συμπεριλάβει ένα μηχανισμό που να σέβεται πληρέστερα τις ισχύουσες ε, δικαιοδοσίες του. Και τελικά ξέρουμε ότι θα υπάρξουν προβλήματα και πρέπει να σεβαστούμε τις συστάσεις του διαμεσολαβητού που ταυτίζουν ένα πραγματικό πρόβλημα για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αν εμείς δεν το καταλάβουμε αυτό στο Κοινοβούλιο, τότε θα σήμαινε αυτό ότι αποφεύγουμε τις πραγματικές μας πολιτικές ευθύνες. Ας δούμε λοιπόν τι τροπολογίες θα κατατεθούν μέχρι αύριο και θα προσπαθήσουμε να τις συμπεριλάβουμε σε συμβιβαστικές για να είναι καλύτερη η έκθεση των δύο επιτεροπών. Ευχαριστούμε κυρία Μετσόλα, η κυρία Κέλλερ. Και εγώ ευχαριστώ όλους και όλες για τα σχόλιά τους. Όπως είπε και η κυρία Μετσόλα προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι πρακτικό και για τους πρόσφυγες και μετανάστες ώστε να μπορούν να διεκπαιρεωθούν τα παράπονά τους Οι λεγόμενοι guest officers είναι στα σύνορα με ειδική λωρίδα στο μανίκι τους που γράφει Frontex, Frontex, Montex. Και ε, έτσι θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να γίνουν ακόμη πιο πρακτικά και να αποτελέσουν μέχρι και πρότυπο. Νομίζω ότι κινούμεθα προς τη σωστή κατεύθυνση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων για το Frontex και για την Ένωση γενικότερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και προσβλέπουμε στις τροπολογίες σας. Ευχαριστούμε η Ακέλερ μου. Η διορία κατάθεση τροπολογιών λήγει αύριο στις 12. Και τώρα Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω το απόγευμα να φέρετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες γιατί θα ψηφίσουμε. Θα ξαναειδωθούμε σε λίγο. Ευχαριστούμε.